Ε, όπως γνωρίζουμε όλοι, η κράτηση είναι διοικητική πράξη. Δεν επιβάλλεται ε, στους εισερχόμενους γιατί έχουν διαπράξει κάποιο ποινικό αδίκημα. Επιβάλλεται για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης διαδικασίας που αποφασίζεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να στερείς την ελευθερία των ανθρώπων για τις ανάγκες της διοίκησης. Είναι πολύ σκληρή η επιλογή της κράτησης σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο επιβάλλεται. Ε, έτσι βλέπουμε πολύ συχνά κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν το θεσμό της κράτησης ως ε, μηχανισμό αποτροπής εισόδου προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή ως φόβητρο να μαθαίνουν οι εισερχόμενοι ότι δεν θα περάσουν καλά σε μια χώρα, θα κρατηθούν ενδεχομένως για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να μην τολμάνε να μπαίνουν στη χώρα για να ζητήσουν ή όχι άσυλο. Ε, αυτό δημιουργεί, ε, όπως καταλαβαίνουμε, προβλήματα στην ελευθερία των ατόμων και στα δικαιώματά τους να ζητάνε άσυλο σε όποια χώρα θεωρούν ότι μπορούν να, προστα... να ζητήσουν διεθνή προστασία. Ε, εκείνο το οποίο λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι μπορεί μερικά άτομα να ε, καταχρηστικά να ζητάνε άσυλο χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις του πρόσφυγα δεν μπορεί όμως τα κράτη-μέλη να απαντούν εξίσου καταχρηστικά και να επιβάλλουν την κράτηση με μάλιστα με διάρκεια που πολύ συχνά είναι υπερβολική διότι σε αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει και είναι δεδομένο ότι ποτέ δεν ευθύνεται ο διοικούμενος για την αδυναμία της διοίκησης να προχωρήσει στην έρευνα ενός αιτήματο ασύλου. Αν λοιπόν η διοίκηση δεν μπορεί να εξετάσει τα αιτήματα ασύλου, δεν μπορεί να αποφασίζει να κρατηθεί ένα ετών άσυλο για περιόριστο χρονικό διάστημα. Επίσης έχει υποθεί και το έχουμε αποδεχτεί, συγγνώμη ένα δευτερόλεπτο, ότι δεν μπορεί να αποφασίζεται κράτηση στις ευάλωτες ομάδες. Καταρχήν στα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει κανένα σκοπός που να προσφέρεται η κράτηση στα παιδιά ή σε άρρωστους ή σε υπερήλικους ή σε ανθρώπους που είναι ανήμποροι να επιβιώσουν σε κέντρα κράτησης. Αυτά λοιπόν τα ζητήματα πρέπει να τα τονίσουμε. Όταν μιλάμε για κράτηση δεν μπορούμε να μην θέσουμε αυτά τα ζητήματα εισαγωγικά και να πούμε ότι η κράτηση είναι μόνο κατεξαίρεση έτσι λέει ο νόμος, έτσι είναι όλη η φιλοσοφία, πρώτα τα εναλλακτικά μέτρα της κράτησης και αν τελειώσουν αυτά και δεν μπορείς να εξασφαλίσεις την παρουσία του πρόσφυγα στη διαδικασία ασύλου, μόνο τότε η κράτησή του και όχι κράτηση σε ευάλωτες ομάδες και όχι κράτηση γιατί η διοίκηση δεν μπορεί να καταφέρει και η υπηρεσία ασύλου να ερευνήσει τα αιτήματα. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Um, as we have a little bit time, I would like to add another question, because first of all, uh, when we talk about legal assistance, I think to